So, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ καθίστε. Για να αρχίσουμε σιγά σιγά τη συνεδρίαση. Καλωσορίζω ε, θερμότατα τα εγγόνια του συναδέλφου Βιτόριου πρώτη. Δύο είναι εδώ πίσω. Καλωσορίζω την αντιπροσωπεία από την Ιταλία. Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που ήρθατε να δείτε τον παππού σας να δουλεύει. Είναι πρέπει να σας πω και από τους πιο επιμέλεις βουλευτές και μπορείτε να είστε περήφανοι για τον παππού σας. Έχουμε και έναν άλλον ιδιαίτερο προσκεκλημένο και θέλω να ε, καλωσορίσω τον Υπουργό ε, Υγείας της Λιθουανίας, τον κύριο ε, Κάιτης και ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε, που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να μας ενημερώσετε και για το ίδιο το πρόγραμμα της Προεδρίας. Είχαμε και μια συνομιλία προηγουμένως και την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σας έχει ιδιαίτερη σημασία για λόγους οικογενειακής ιστορίας αλλά και για το μέλλον πρέπει να πω. Ε, για την πολιτική υγεία. έχουμε ορισμένα πράγματα εδώ να εκκρεμούν, ορισμένα θέματα υγεία. Βλέπω εδώ την Dagmar μπροστά μου ε, που έχει την έκθεση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, medical devices και κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα έχουμε να συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται να μακρηγορώ εγώ. Σας καλωσορίζω θερμότατα. ήρθε και ο Υπουργός Γεωργίας ε, και ε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ε, τώρα έχουμε τον Υπουργό Υγείας. Έχετε το λόγο για τις προγραμματικές δηλώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμε πρόεδρε της Επιτροπής, περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα τη Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Στα γερμανικά. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, όσο και μεγάλη ευθύνη, η ευκαιρία που έχω να σας παρουσιάσω ε, το πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας για την Υγεία. Πριν από λίγες μέρες μόλις είχα την τιμή να ε, προεδρεύσω στην άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Υγείας στο Βίλνιος όπου και τους υποδέχτηκα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εφήγησαν πάρα πολύ σημαντικά θέματα υγείας για όλα τα κράτη-μέλη. Όπως είναι η βιωσιμότητα και η των συστημάτων υγείας, η ψυχική υγεία, ε, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, η κατανάλωση ε, προϊόντων καπνού από τους νέους. Είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ε, έχουν εργαστεί από κοινού και έχουν διαμορφώσει και κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας για την οδηγία για τον καπνό. Αυτό είναι μια μικρή αφετηρία. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την πολιτική βούληση η κοινή ε, δράση και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας και σε όλα τα θέματα που άπτονται τη δυσυχία νομίζω θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στην ολοκλήρωση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Όλα τα κράτη-μέλη ελπίζουν κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας να επιτευχθούν μεγάλες πρόοδοι και σε άλλους τομείς όπως είναι τα κλινικά πειράματα, ε, τα ιατρικά σκευάσματα ή τα τέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ιδιαίτερα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διαμορφώσουμε ενιαία άποψη στο Συμβούλιο Υπουργών και κοινή θέση, για παράδειγμα, ε, στις ιατρικές δοκιμές. Αυτό θα πρέπει να προχωρήσει με πιο ε, γρήγορους ρυθμούς και να εξασφαλίσει και την πρόοδο και άλλων θεμάτων. Σήμερα στην Επιτροπή σας έρχομαι να σας μιλήσω και ε, ε, αισθάνομαι θετική ενέργεια από το Συμβούλιο και πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα συνεργασίας εδώ και πραγματικά ε, είναι μεγάλη η συνεργασία μας και η αισιοδοξία. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα αγγλικά. Θα σας πω γιατί αισθάνομαι συγκίνηση. κατά τη διάρκεια της Προεδρίας ξέρετε ότι η κατάσταση και η σύνθεση της ε, νομοθετικής δομής είναι γνωστή σας σε εξαιρετικό τρόπο και δεν είναι η πρώτη φορά που ακούει κανείς τα λόγια ο στόχος μας μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα λόγια ωστόσο είναι δοκιμασμένα από τη ζωή και για τη Λιθουανία το ίδιο. Πήραμε την Προεδρία από την Ιρλανδία και είμαστε η πρώτη χώρα που έχει αυτή την ε, βαλτική χώρα που έχει αυτή την ευθύνη. Τα λόγια αυτά δοκιμάστηκαν μια φορά για όλα. Η Λιθουανία, η Λετωνία και η Εστονία. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα γκουλάγ στη Σιβηρία. Ανήκα στο κίνημα των αντιφρονούντων της Λιθουανίας και ήξερα τι σημαίνει για μένα και για τους συντρόφους μου η έγκριση στις 13 Ιανουαρίου του 1983 ενός ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση στις βαλτικές χώρες που υποστήριζε την ελευθερία των χωρών αυτών. Το Κοινοβούλιο απάντησε στο αίτημα 45 αντιφρονούντων των βαλτικών χωρών προς το δημοκρατικό κόσμο, ζητώντας την, ε, τις, ε, ε, τονίζοντας τις επιπτώσεις και την ανάγκη διάλυσης του συμφώνου Ρίτεντροπ Το... Αυτό έδειξε ακριβώς το alle Menschen Brunnen. Όλοι, όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια. Επιτρέψτε μου λοιπόν Μάτιας. On this occasion... Κύριε Πρόεδρε, με την ευκαιρία αυτή να σας δώσω ένα βιβλίο για την σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας στείλω σε όλους σας ένα αντίτυπο. Ευχαριστώ και τονίζω ότι μόνο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρήσουμε και την βασική έννοια και την ευρωπαϊκή και την θετική προοπτική της ε, Ευρώπης. Ο Γιούστας Παλέσκας, ο οποίος ήταν ένα μέλος του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας τον καιρό της Ανεξαρτησίας και παρόν εδώ τώρα, τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μοναδικό όργανο που εκλέγεται από όλους τους Ευρωπαίους και τους εκπροσωπεί όλους. Το πεπρωμένο με έκανε να γίνω μέλος της συνέλευσης που ετοίμασε το σχέδιο συνθήκης για το Σύνταγμα της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έδωσε σε όλους εμάς την ευκαιρία να δουλέψουμε εδώ στο κτίριο αυτό και να αισθανόμαστε να είμαστε στο σπίτι μας. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην συνέλευση αυτή υποστήριξαν με θάρρος στην αρχή περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη Ευρώπη και έφεσαν ε, και τόνισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα στέρεο σύνταγμα και αποτελεσματικούς μηχανισμούς που θα επέτρεπαν την επίλυση των πιο ευάλωτων, των πιο τροτών ζητημάτων όπως της υγείας. Άλλωστε η αρχή των υψηλότερων δυνατών δικτών υγείας που ενσωματώνει απόλυτα η συνθήκη της Λισαβόνας προήλθε από το σχέδιο, συνθήκης, σχέδιο συνταγματικής συνθήκης της Ευρώπης. Στην Επιτροπή σας λοιπόν μιλώντας ενώπιόν σας, ξέρω πολύ καλά πόσο τεράστια σημασία έχει να δουλεύουμε σαν εταίροι για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Τα επιτεύγματά σας μαζί με την Ιρλανδική Προεδρία στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, την κοινή μεταρρύθμιση της Γεωργίας και της Αλίας, το Erasmus Sin, το, το Life Sin, του κόσμου τα πράγματα μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε για να κρατήσουμε αυτή την θετική και δυναμική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις επόμενες εκλογές, το Μάιο του 2014, θα μπορέσει να εφαρμόσει τις πενταετούς διάρκειες δεσμεύσεις της παρουσιάζοντας τις ενώπιον των λαών της Ευρώπης, ε, προστατεύοντας την ευημερία των Ευρωπαίων και τονίζοντας την ανάγκη να είναι δραστήριοι στις επόμενες ευρωεκλογές. Να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα Η προτεραιότητα της Λιθουανικής Προεδρίας ε, στον τομέα της υγείας είναι να εγκριθεί και να επιβεβαιωθεί η απόφαση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για ε, τα αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα υγείας. Ε, υγεία με την ευρεία έννοια και βιώσιμα θα πρέπει να είναι και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά και όχι μόνο υπηρεσίες υγείας, μιλώ συνολικά για ένα σύστημα υγείας. Είναι σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη, ακόμα και για την ε, οικονομική και την καινοτομία. Γι' αυτό στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο συμπεριλαμβάνονται και μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας. Γι' αυτό χρειάζεται και την απαραίτητη ε, οικονομική υποστήριξη αυτός ο κλάδος τα συστήματα υγείας και η σχετική πολιτική είναι κάτι το καινοφανές ως ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Αυτό δεν θα πρέπει να αφιστούμε κόπων και ε, προσπαθειών ε, για να δώσουμε νέες προοπτικές στους πολίτες της Ένωσης. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων ε, οδηγεί και σε καλά αποτελέσματα και είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Σας καλώ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σας προσκαλώ στο φόρουμ ε, της Υγείας στο Βίλνιου στις 19 και 20 Νοεμβρίου για την αηφόρο και βιώσιμη υγεία σε μια ε, βιώσιμη και αηφόρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα συζητήσουμε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά και τη διασυνοριακή συνεργασία. Είναι μια καλή πλατφόρμα για τη συζήτησή μας. Φέτος λίγη η ευρωπαϊκή στρατηγική υγείας, γι' αυτό θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες στρατηγικές, νέες μεθόδους και μέσα, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή πολιτική υγείας να ενισχυθεί και να προχωρήσει και να συνεχίζει η ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση με τρόπο πιο αξιόπιστο η Προεδρία συνεργάζεται στο τρίο με την προηγούμενη και την επόμενη Προεδρία και μαζί σας ε, επίσης θα εξασφαλίσουμε μια συνέχεια ε, στα σημαντικότερα ζητήματα που άπτονται του τομέα της υγείας. Παράδειγμα, τα κλινικά πειράματα και δοκιμές, τα ανθρώπινα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συσκευές και για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Υπάρχουν όμως ιδιαίτερα κίνδυνοι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό θα πρέπει μεταξύ μας να συντονίζουμε πάντα τη δράση μας. Και παγκοσμίω ε, ε, να συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους άλλους εταίρους της. Αυτό πώς εκφράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση θα... Ε, πρέπει να σας πω ότι κύρωσε τη συμφωνία πλαίσιο του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει πλέον τώρα στην ε, υλοποίηση αυτής της σύμβασης. Τα ίδια ισχύουν και για τον καπνό και την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο να αποφανθεί επίκειται ακόμα αυτή η απόφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι για την υγεία και θα πρέπει να περιοριστεί ε, η κατανάλωση προϊόντων καπνού. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι πολίτες και οι ψηφοφόροι υποστηρίζουν αυτή την πρόταση και αυτή η πρωτοβουλία. Και η χτεσινή ψηφοφορία εδώ το απέδειξε. Ήταν εξαιρετική η ψηφοφορία στην Επιτροπή σας και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, καθώς επίσης και την εισηγήτρια την κυρία Λίντα Μακάβαν. Σας ευχαριστώ πολύ για την αφοσίωσή σας ε, ε, στα θέματα υγείας των πολιτών και ελπίζω σε συνεργασία με τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ματίας Γκρότε και την ε, κυρία Λίντα Μακάβαν, την Γλένις Βίλμο, την Ντάγμα Λοτ Μπέρεντ, τον Πέτερ Λίζε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για αυτά τα θέματα. Όλα τα ιατρικά ζητήματα, όλα τα ζητήματα υγείας να τα φέρουμε σε αίσιο πέρας. Είμαι στη διάθεσή σας. Έχω κάθε προεθυμία και κάθε καλή θέληση να σας ακούσω, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσω τις προτάσεις σας. Και στο πνεύμα του διαλόγου ε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εργαστώ με πολύ μεγάλη ευθύνη ε, και ζήλο το επόμενο εξάμηνο. Ποιο εξάμεινο, τετράμινο ουσιαστικά είναι για τις εργασίες μας. σε λίγο θα πάτε στις διακοπές σας που τις χρειάζεστε γιατί πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας ε, το επόμενο εξάμεινο, ιδιαίτερα στην προεκλογική εκστρατεία για να είστε υγιείς ε, και με σφρίγος να αντιμετωπίσετε ε, την προεκλογική εκστρατεία. Αλλά προηγουμένως το φθινόπωρο θα χρειαστεί να συνεργαστούμε μαζί για τα θέματά μας και είμαι πεπισμένος ότι και τα 28 κρατα ημελη έχουν καταλάβει στο άτυπο συμβούλιο πόσο αποφασιστική είναι αυτή η περίοδος. Διότι το επόμενο έτος θα ανοίξει νέες προοπτικές και νέα δεδομένα θα φέρει. Τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να τα προωθήσουμε και να ολοκληρωθούν. Σας είπα ποια είναι τα ζητήματα, οι κλινικές δοκιμές, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Εγώ δεν μπορώ να τα πετύχω μόνος μου. Χρειάζομαι την υποστήριξη της Επιτροπή σας με επίσημες και άτυπες επαφές και συναντήσεις. Σας ευχαριστώ και περιμένω με ενδιαφέρον τις ερωτήσεις. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι πρόεδρος από το Γενάρη του 2012, αλλά Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από αυτό που άκουσα τώρα μόλις. Όχι μόνο για τα θέματα επί της ουσίας που μας παρουσιάσατε, που επίκυνται, αλλά και μας είπατε και την προσωπική σας ιστορία και πώς είστε συνδεδεμένος με την Ευρώπη και ποια ιδέα έχετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δεν είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά και μια συναρπαστική υπόθεση. Και δεν είναι μόνο ένα ιστορικό εγχείρημα, αλλά και ένα εγχείρημα για το μέλλον και για την υγεία Νομίζω πολύ ωραία τα είπατε. Σπάνια έχω ζήσει μια τέτοια ε, ομιλία. Με εντυπωσιάσετε. Ευχαριστώ για το βιβλίο. Θα το διαβάσω στις διακοπές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας μπούμε τώρα στη συζήτηση. Πρώτα οι συντονιστές και ο Πέτερ Λίζε που είναι συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, για θέματα υγείας. Στη συνέχεια η συνάδελφος Λίντα Μακ Άβαν. Ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πραγματικά πρέπει να σας πω, ήταν πάρα πολύ ζωντανή η παρουσίασή σας, πάρα πολύ ζωηρή. Έχετε την απαραίτητη ενέργεια ε, για να προωθήσετε τα ζητήματα υγείας. Για τα προϊόντα καπνού το Συμβούλιο έχει προχωρήσει αρκετά. Τώρα το θέμα είναι να βρεθεί συμφωνία με το Κοινοβούλιο γιατί εκκρεμούν και άλλα σημαντικά ζητήματα, τα ιατρικά προϊόντα, ε, ε, τα, οι κλινικές δοκιμές και ε, in vitro το Συμβούλιο δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει μια συμφωνία και εμεί θέλουμε να πούμε στους συναδέλφους σας ότι χρειάζεται να δράσουμε. Του χρόνου έχουμε ευρωεκλογέ και ουσιαστικά μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο θα πρέπει να έχουμε καταλήξει για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια πριν τι εκλογές. Οι πολίτες στην Ευρώπη θέλουν καλύτερη προστασία της υγείας τους και πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ζητώ εδώ επίσημα να απευθανθείτε ε, στους συναδέλφους σας και στις υπηρεσίες του Συμβουλίου, τους υπαλλήλους, για να προωθηθούν αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε το αργότερο Οκτώβριο-Νοέμβριο να πάμε στους τριμερείς διαλόγους. Δεν γίνεται πια. Ε, στη δική μου έκθεση, ε, τη διαγνωστικές μεθόδους in vitro, θα ήθελα να σας πω τι συζητήσαμε με τους σκιώδεις ηγητές και τους άλλους συναδέλφους. Και που το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μια ρύθμιση για ε, την ενημερωμένη συνένεση στις γενετικές δοκιμές, δηλαδή να ενημερώνονται οι ε, πολίτες γιατί έχει δραματικές συνέπειες ε, αυτή η ιστορία και μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορεί να τους συμβουλεύουν έτσι εμπορικά και εμπαρόδορισμένοι. Χρειάζονται γιατροί με επαγγελματισμό, με πλαισίωση. Δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά την αρχή ε, πραγματικά ναι. Για τα τρία θέματα που σας ανέφερα, κλινικές δοκιμές, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι βίτρο διαγνωστικές μέθοδοι, ε, θα ήθελε το Κοινοβούλιο να βάλει το ρόλο της, της Επιτροπής ε, στα κείμενα, που δεν υπάρχει σήμερα στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, θέλουμε ο συμβασμός να αναγράφει ε, συμφωνία, η σύμφωνη γνώμη μιας ε, τέτοιας επιτροπής. Αυτό το λέει η δήλωση του Ελσίνκη και εσείς είστε και γιατρός και γνωρίζετε τι σημασία έχει η διακήρυξη του Ελσίνκη παγκοσμίω για τους γιατρούς και προσβλέπω και ελπίζω στη συνεργασία σας έτσι ώστε όλα αυτά να κατοχυρωθούν και στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ισχύει και σήμερα. Ένα τελευταίο. Στην οδηγία για τις κλινικές δοκιμές, τα πειράματα, σήμερα απαγορεύεται ακόμα ε, η ε, ε, επέμβαση στο, στα πλαστικά κύτταρα, τα ανθρώπινα. Αποφάσισε η Επιτροπή μας με μεγάλη πλειοψηφία να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Μια που είστε και γιατρός λοιπόν, παρακαλώ φροντίστε να υιοθετήσει ε, αυτή την τροπολογία του Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Μακάβαν που δεν είναι μόνο συντονίστρια των σοσιαλιστών και δημοκρατών, αλλά και η συγγήτρια, όπως γνωρίζετε, για τα προϊόντα καπνού και την αντίστοιχη οδηγία, αλλά και η συγγήτρια για την φάρμακο επαγρύπνηση και από σήμερα για ένα τρίτο θέμα. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργέ, πραγματικά με ικανοποίησαν αυτά που άκουσα. Ε, δεν είμαστε σε αισιόδοξο στάδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλό είναι να θυμίζουμε την ιστορία της γυραιάς Υπήρου, να θυμόμαστε ότι ζούμε μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη και για πρώτη φορά στην ιστορία μας από την ε, Ιρλανδία μέχρι τα σύνορα με τη Ρωσία έχουμε δημοκρατικά καθεστώτα. Είναι μεγάλο επίτευγμα και τίνουμε να το ξεχνούμε λόγω απεσιοδοξίας. Πραγματικά είναι καταπληκτικό που μας το θυμήσατε και ας ε, το σκεφτούμε και τη διάρκεια των διακοπών μας εν ώψη των εκλογών η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέκτησε κάτι πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και σημαντικό το μήνυμά σας. Θα επιστρέψω τώρα στην καθημερινότητα των εργασιών μας. Ε, ξέρετε ότι ε, κατηδίαν συζητήσαμε και για τη χθεσινή ψηφοφορία για τον καπνό και χαίρομαι με τη δέσμευση που έχετε αναλάβει, δηλαδή ε, συμφωνία προτού λήξει η Προεδρία Υπάρχει κοινή θέση του Συμβουλίου για τη σχετική οδηγία. Εμείς το Σεπτέμβρη θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και ευελπιστώ ότι με το που ψηφίσει το Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να έχουμε και μια θετική έκβαση για να προωθήσουμε ε, την δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με τις ε, κλινικές δοκιμές και αυτά που είπε ο Πίτερ Λίζε ε, και είχαμε πριν από δύο μήνες, ε, ε, μία ψηφοφορία στην Επιτροπή ήταν σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη. Θέλουμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, διότι χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία για τις κλινικές δοκιμές, ε, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά για να συνεχιστεί και η έρευνα στην Ευρώπη και να παραμείνει θέση απασχόλησης όσο έχουν για τις κλινικές δοκιμές στον ερευνητικό τομέα της Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν να σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, αν μπορείτε να επεκταθείτε λίγο. Και κάτι άλλο, οι αμοιβέ τα τέλη, συγγνώμη για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Ήμουνα εισηγήτρια για το βασικό νομοθέτημα πριν από δύο χρόνια και ελπίζω να ε, ταχύτατα να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε, Λίντα. Ε, κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ήταν εντυπωσιακή. Είδαμε και αν είδαμε υπουργού από την αρχή της Προεδρίας σας, αλλά αξίζεται την ιδιαίτερη προσοχή μας. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όχι μόνο για το θεματολόγιο σας, αλλά και για τα βιώματά σας που μας μεταφέρατε. Ε, είμαι η συγγήτρια για ένα ε, δύσκολο φάκελο ναι, και αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις ε, τη διάρκεια της Κυπριακής ε, Προεδρίας. Η Ιρλανδική Προεδρία μας βοήθησε πάρα πολύ, ήταν πολύ αφοσιωμένη, αλλά όλοι οι αρμόδιοι για αυτό το ζήτημα, αλλά το Κοινοβούλιο κατέβαλε επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσει να πλησιάσει το Συμβούλιο ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξάλλου σε μεγάλο βαθμό τροποποίησε την αρχική της πρόταση και ευθυγραμμίστηκε με την θέση του Κοινοβουλίου. Δεν βλέπουμε όμως ε, να γίνονται βήματα για να απεμπλακεί ο φάκελος στο Συμβούλιο προχωρούν όλα πολύ αργά και ναι. στα μάτια της κοινή γνώμης ε, με αυτή την νομοθεσία θα μπορέσουν όλες οι εθνικές αρχές αλλά και οι πολίτες να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, να υπάρχει διαφάνεια για τιμολόγηση των φαρμάκων αλλά κυρίως για την αποζημίωση των φαρμακευτικών ταπανών. Για τη Λιθωνική Προεδρία ελπίζουμε αυτό να αναδειχθεί ε, σε προτεραιότητα και βασιζόμαστε στη μελλοντική σας υποστήριξη. Ποια είναι δε η γνώμη σας, πώς μπορούμε να τονώσουμε λίγο την όλη διαδικασία και κυρίως στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε. Ο Κάρις Σλίτερ τώρα. Ευχαριστώ που ήρθατε, Υπουργέ. Καλωσορίζω το ότι ρητά αναφερθήκατε στην σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού. Α, είμαι σε λάθος μικρόφωνο. Αυτό θα πρέπει να καθοδηγήσει τις εργασίες μας. Είναι αυστηρός ο κανονισμός σε σχέση με τις επαφές με τα λόμπι και αυστηρούς κανόνες για τη δημοσίευση πληροφοριών και τη διαφάνεια. Ε, αναρωτιόμουν ε, με ποιο τρόπο θα πείσετε τους συναδέλφους σας να συμμορφωθούν ε, με αυτές τις αυστηρές διατάξεις. Θέλουμε να επιτύχουμε πλήρη διαφάνεια και στο Συμβούλιο κατά την επεξεργασία του φακέλου των προϊόντων του καπνού. Ε, Χθε στην Επιτροπή είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Το 75% της υποστήριξη είχαμε στην Επιτροπή. Υποστηρίζουν το 65% γιατί κάποιες χώρες δεν δέχονται το 75% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μπορούμε να κάνουμε για να υπερπηδήσουμε αυτές τις διαφορές. Υπάρχει και άλλη μια επιχειρηματολογία να μην δεχτούμε την απαγόρευση για τα ε, προϊόντα slim, ε, τα τσιγάρα slim. Ε, για τη διαφάνεια τώρα είναι στοιχείο κλειδί. Ε, έχουμε ιστορικά δεδομένα βάσει των οποίων ε, η έλλειψη πρόσβαση στις μελέτες για τις κλινικές δοκιμές ε, συνεπάγεται ότι οι παρενέργειες που θα μπορούσαμε να έχουμε εντοπίσει μέσω των μελετών τελικά δεν εντοπίστηκαν διότι είναι απόρριτες οι πληροφορίες των μελετών. Λοιπόν, τι πιστεύει το Συμβούλιο για το απόρριτο των μελετών για τις κλινικές δοκιμές. Τελευταία ερώτηση για το αλκοόλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη σκέψεις της για την ε, στρατηγική σε αυτό το τομέα. Τι προβλέπετε για την Προεδρία σας, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες ε, του χρόνου, θα λάβουμε δε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, σήμανση των προϊόντων που δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοθέτημα για τις πληροφορίες σχετικά για τα τρόφιμα και ως υπουργό Υγείας δεν είστε άμεσα αρμόδιος, αλλά σίγουρα θα ενδιαφερθείτε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, για ένα Ρόσμπα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα. Λίγοι είμαστε σήμερα, Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Αλλά κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε και ξανα, να μα ξανάρθετε όταν έχουμε πολύ κόσμο. Θέλω να σα παρουσιάσω, να σα ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, πολύ ζωντανή παρουσίαση που μα κάνετε φυματίωση. Ένα θέμα που θέλω να σχολιάσω. Παραμένει απειλή σε όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς είναι ένα θέμα που δεν το προσέχει ο κόσμος. Ωστόσο, κάθε ώρα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη πεθαίνουν 7 άτομα από φυματίωση. Δύσκολα μπορεί να το καταλάβει, να το δεχτεί κανείς. Πέντε χώρες της Ένωσης ανήκουν στις πλέον θυγόμενες χώρες με βάση τον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό επιτυχίας της θεραπείας της ε, φυματίωσης, πιο πιθανό είναι να θεραπευτεί στο Κονγκό παρά στη Ρουμανία. Το ποσοστό θεραπείας στο Κονγκό είναι 50% και στη Ρουμανία 20%. Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών ούτε καν ξέρουν ότι έχουν φυματίωση. Δεν έχει γίνει διάγνωση. Πάνε στο ίντερνετ, παίρνουν διάφορα φάρμακα που βρίσκουν έτσι και πολύ αργά, πολύ αργά καταφέρνουν να πηγαίνουν σε ένα γιατρό. Πρόκειται λοιπόν για ένα σοβαρό πρόβλημα που εξελίσσεται. Σας είχα στείλει μία επιστολή τέλη Μαΐου, δεν μου απαντήσετε, γι' αυτό θέλω το θέμα ενώπιον σας ελπίζω να, είναι, να, υπα, να, την Προεδρία και το Υπουργείο σας. Και θα ήθελα το θέμα αυτό να περιλαμβάνεται στις ε, προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Σε συνέχεια αυτό που είπα, πιστεύω ότι η πολυανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που συνδέεται άλλωστε και με τη φυματίωση. Γιατί διαπιστώνουμε ότι λόγω του ότι ε, παίρνουμε πολλά φάρμακα, μειώνεται η δυνατότητα θεραπείας της φυματίωσης. Η αντοχή δηλαδή στα αντιβιωτικά αυξάνεται. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι, θα κάνετε προτεραιότητα το θέμα αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό για το πρόβλημα της υγείας στην Ένωση. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εξετάσουμε βέλτιστες πρακτικές, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο, γιατί πολλά μπορεί να μάθει ο ένας από τον άλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιούστα Παλέτσκης, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, στην παρουσίασή σας. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε και πολύ ωραία. Και θέλω να πω και στους συναδέλφους ότι είστε ο πιο δημοφιλής υπουργό στη Λιθουανία. Και ακριβώς είστε τόσο δημοφιλής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, γιατί δεν περιορίζεστε στα λόγια, αλλά περνάτε και στα έργα. Κάνατε τη μεταρρύθμιση της υγείας στην Λιθουανία και ε, προσπαθείτε να εξασφαλίσετε πρόσβαση στην υγεία και για τους πιο απόρους και για τους πιο φτωχούς. Βεβαίως, σας επικρίνουν κιόλα. Αλλή Δεν ε, υπάρχει ε, στην Ευρώπη σήμερα κοινή πολιτική υγείας, αλλά Θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, τι μπορεί να κάνει η Λιθουανία για να φτάνει η, ε, παροχή υγείας και στους πιο πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί να βοηθήσει η Λιθουανία προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα. Στη Λιθουανία Έχουμε πολλούς καλούς γιατρούς ε, οι οποίοι φεύγουν και από άλλες ανατολικές χώρες ε, προς τη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε αυτό το πρόβλημα διαρροής εγκεφάλων και γιατρών. Πώς μπορείτε να το λύσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριος Πρόντι. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας και για την μαρτυρία σας υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου που αντλήσατε και από την προσωπική σας προσωπική αλλά και εθνική ε, ζωή. Εγώ σέβομαι και τη θέση σας και με, μου δίνει ε, βεβαιότητα διότι στηρίζεται στο ότι ένα άτομο μπορεί να δράσει υπέρ της αξιοπρέπειας του καθενός μας. Και αυτό είναι κάτι που εγώ πάντα το τονίζω, γιατί πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Θέλω επίσης να δώσω έμφαση, να υπογραμμίσω την έμφαση που δώσετε στην ψυχική υγεία, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα κεφάλαια μιας προσωπικής αδυναμίας του ατόμου, που πρέπει να υποστηριχθεί και από το υγειονομικό σύστημα, ιδίως όμως από ένα δεκτικό κοινωνικό πλαίσιο. Όλο αυτό το συνολικό πρόβλημα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε συστημικά, σαν ένα σύστημα. Εκτίμησε ιδίως την έμφαση που δώσετε στον καπνό και σε όλη την πολιτική μείωση ε, του κινδύνου που συνδέεται με την πρόσληψη νικοτίνης που αποκλείει τον καπνό. Θέλω να υπογραμμίσω ότι φοβάμαι πως το, το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να αποτελέσει πιο ευέλικτο εργαλείο ε, πρόσληψης βαρέων ναρκωτικών, διότι μία εισπνοή ε, ισοδυναμεί με εισπνοή ε, δηλητηρίου. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος το που με ε, ε, θα ήταν κάτι λοιπόν που πρέπει να εξετάσουμε. Δεν θα πρέπει ε, να χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο σαν ε, για να παρέχεται ε, με άλλο τρόπο ένα επικίνδυνο ναρκωτικό. Θα περιοριστώ λοιπόν στην ανάγκη να υπογραμμίσω εκ νέου το πρόβλημα που έφεσαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ πήρατε τόσα μπράβο που και εγώ συμφωνώ βεβαίως μαζί σας, δεν θα σας πω άλλα μπράβο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον που σας ακούσαμε, όπως και κάποιους από τους συναδέλφους σας, διότι εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Εντάξει, πολύ φιλόδοξα όλα αυτά που μας λέτε και πάρα πολύ αξιέπαινα, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι στο υπόλοιπο του έτους που είναι 4,5 μήνες ως πραγματικός χρόνος εργασίας, οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Γι' αυτό μου αρέσει ε, που θέτετε προτεραιότητες και έχω και πολλά θέματα που δεν είναι ε, νομοθετικού περιεχομένου, ε, δεν θα τα αναφέρω. Είδα ότι ασχολείστε με την ψυχική υγεία και κάνετε και αντίστοιχη διάσκεψη, πολύ σπουδαίο αυτό και για τα υπόλοιπα θα παρακαλούσα να περιοριστείτε να τηρήσετε τα νομοθετικά. Κοίταξα το κείμενό σας και βλέπω πώς περιγράφετε την πρόοδο που θέλετε να επιτελέσετε. Ξέρετε, αυτό με οδήγησε σε μηδίαμα λίγο, γιατί ε, είδα μια κάποια ειλικρίνεια και μ' αρέσει αυτό. Λέτε ε, για τον καπνό τίποτα. Άρα θεωρείτε ότι θα είναι δύσκολο να βρείτε ένα αποτέλεσμα. Για τις κλινικές δοκιμές λέτε ότι επιθυμείτε σημαντική πρόοδο, significant progress. Και επίσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που με ενδιαφέρει εμένα, γράφετε ότι πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί καλή πρόοδος Είναι σημαντική διαφορά για τα διάφορα θέματα, το πώς αξιολογείτε την πρόοδο που μπορείτε να ε, πετύχετε. Γι' αυτό θα ήθελα να μου δώσετε μια πολύ ειλικρινή απάντηση παρακαλώ. Τι πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει η ομάδα εργασίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Εγώ περίπου έχω μια ιδέα. Με ποια από τα άρθρα μέχρι τώρα έχει ασχοληθεί αυτή η ομάδα εργασίας. Εσείς πιστεύετε ότι μέχρι τα τέλη του έτους, άντε Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα έχουμε πραγματικά μπει σε εντατικούς τριμερείς διαλόγους για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με εσάς. Γνωρίζετε ότι και αυτά που λέει ο κύριος Λίζα και αυτά που λέω εγώ έχουν να κάνουν μεγάλη σχέση με την ασφάλεια των ασθενών. Και δεν είμαι καθόλου αφελής για να σας ρωτήσω ποια μορφή εμπορίας αυτών των τεχνολογικών προϊόντων υποστηρίζετε. Δεν θα μου το πείτε. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν πρώτερη έγκριση ή να ενισχύσετε τους οργανισμούς κοινοποίηση. Το ξέρω ότι δεν θα μου το απαντήσετε, γι' αυτό δεν σας το ρωτάω κιόλα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να μάθω παρακαλώ, γιατί με ενδιαφέρει, είναι το χρονοδιάγραμμά σας πότε περίπου να περιμένουμε να μπορούμε να συζητήσουμε για λεπτομέρειες. Και εγώ και ο κύριος Λίζα για τις εκθέσεις μας. Μπορούμε να συζητήσουμε με την επικεφαλής της ομάδας εργασίας για λεπτομέρειες άρθρο-άρθρο. Εκεί θα παρακαλούσα μια σαφή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ροτ Μπέρεντς. Άλλους δύο έχουμε τώρα. Η κυρία Μαρκουνάιτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω θερμότατα εδώ στην Επιτροπή μας. Ήταν πολύ ωραία η παρουσίασή σας πραγματικά και σας ευχαριστώ για τις προτεραιότητες που μας αναφέρατε. Θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω το συνάδελφό μου, το Λιθουανό, για την μεταρρύθμιση της υγείας στη Λιθουανία. Βεβαίως υπάρχουν και επικριτικές φωνές που ακούγονται και δεν ξέρω αν καταφέρετε πραγματικά εσείς να λύσετε τα προβλήματα. Εάν θέλετε να καταργήσετε τον ιδιωτικό τομέα από τις υπηρεσίες ε, παροχής υγείας. Πολύ συχνά Προσπαθούμε εμείς εδώ να λύνουμε προβλήματα, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Και ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να ενημερώνεται καλύτερα ο κόσμος ε, για τις ουσίες και για τα προϊόντα που βλάπτουν την υγεία του. Δεν ξέρω, ίσως κάποια ενημερωτικά προγράμματα από παιδική ηλικία, από τα σχολεία, για να γνωρίζουν και οι νέοι μας και τα παιδιά τι είναι καλό και τι είναι κακό για την υγεία. Άλλο πρόβλημα είναι η νόσοι που πλήττουν το γυραιότερο πληθυσμό, ε, τύπου Alzheimer κλπ. Και αυτό το συζητούν στο πρόγραμμα Horizon 2020, μήπως θα μπορούσατε να αναφερθείτε και σε αυτό το πρόβλημα και να μας πείτε ε, ποιες είναι οι προθέσεις του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Η νέα συνάδελφος από τη νέα χώρα, μέλος στην Κροατία. Ε, είναι παρθενική ομιλία σας και όλα στην Επιτροπή μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Η συνάδελφος Πόλσα. Ε, Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω διότι πρέπει να τα είπατε πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ και εγώ για την δουλειά που κάνετε. Είχαμε συναντηθεί στο Ζάγκρεμπ. Θέλω να τονίσω κάτι που μας ενδιαφέρει δύο στην Κροατία και ενδιαφέρει και το κοινό. Ερώτημα που συχνά τίθεται. Με την προσχώρηση της Κροατίας στην Ένωση υπάρχει ο φόβος ότι θα υπάρξει έξοδος του ιατρικού προσωπικού κυρίως των νοσοκόμων δηλαδή, προς άλλες χώρες της Ευρώπης. Η κρίση ε, μας φοβίζει και καταλαβαίνετε ότι φοβίζει και αυτούς. Είχατε την ίδια κατάσταση, αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα στην ε, Λιθουανία. Μετά, το πρόγραμμα δράσης e-health, το δίκτυο δηλαδή δημοσίων οργανισμών υγείας της Ευρώπης που προχώρησε σημαντικά. Ιδίω χάρη στα μέτρα που λέφθηκαν το 2008. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρει αυτή η δυνατότητα για να μειωθεί και το κόστος των ε, ιατρικών δαπανών. Η, η εξέλιξη των τεχνολογιών έχει επίπτωση και στις ιατρικές τεχνολογίες, ωστόσο οι εξελίξεις αυτές ούτε παρακολουθούνται συστηματικά, ούτε ρυθμίζονται συστηματικά. Γι' αυτό χρειάζεται μία ταχύρυθμη διαδικασία προσαρμογής τους στις νέες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος ε, των ομιλητών. Έχει το λόγο ο Υπουργό για να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δώσει και ίσως και κάποιες νέες σκέψεις σχόλια. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Κανονικά θα πρέπει να απαντήσω σε λεπτομέρειες σε κάθε ερώτημα σας, γιατί πραγματικά είστε ε, πάρα πολύ ειλικρινείς και ρωτάτε με ανοιχτό πνεύμα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα αρχίσω από τον Πέτερ Λίζε, με τον οποίο συναντήθηκα προλίγου. Αυτό που με ρώτησε συνδέεται και με την ερώτηση της κυρίας Ροτ Μπέρεντ και γενικότερα με το τρί πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε αυτό το τετράμινο να το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα και να έχουμε αποτελέσματα. Συνεδρίασε ένα άτυπο συμβούλιο και πιστέψτε με ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης εξέφρασαν την εξής ε, επιθυμία οι υπουργοί. Είπαν Κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας έγινε μια πρώτη προσπάθεια. Δημιουργήθηκε μια κοινή αφετηρία. Τώρα είστε το ερώτημα ε, ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Λιθουανίας. Τι καινούριο θα κάνει, τι επιπλέον θα φέρει εμείς είπαμε ότι αν υπάρχει βούληση ε, από τις 28 χώρες θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα ε, καταλήξουμε. Ε, το in vitro, τις διαγνωστικές μεθόδους, τα ιατροτεχνολογικά ή τις κλινικές δοκιμές. Αυτά τα τρία έχουμε. Ας απαντήσουμε ειλικρινά. Ποιο θέμα από αυτά μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Για τις κλινικές δοκιμές τα επίμαχα σημεία δεν είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε, εφόσον λυθούν βεβαίως τα τεχνικά ζητήματα. Ε, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υπάρχουν ακόμα πολλά τεχνικά ζητήματα να ξεκαθαριστούν. Το κοινοβούλιο όμως, ομόφωνα περίπου, ε, έχει εκπονήσει μια θέση ενιαία. Το Συμβούλιο είναι εκείνο που καθυστερεί. Ε, στη συζήτηση λοιπόν με τον Πέτερ Λίζε είπα ότι ας αρχίσουμε από την ημερήσια διάταξη της ομάδας εργασίας και εσείς οι βουλευτές έχετε άμεση επαφή με τις κυβερνήσεις σας. Απευθυνθείτε στις κυβερνήσεις και αξιοποιήστε και τους επίσημους διάβλους και τους άτυπους. Εγώ είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους μου και τους 27 και να τους πω ότι χρειαζόμαστε μια καμπή τώρα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Μιλώ πάντα για τις κλινικές δοκιμές και τα πειράματα. Είναι καλό και σημαντικό και για τους ασθενείς και για την έρευνα και για την επιστήμη και για την καινοτομία και για τις επενδύσεις. και για να παραμείνει όπως οφείλει ανταγωνιστική Ευρώπη. Όλα αυτά είναι επίκαιρα προβλήματα και μας αφορούν όλους. Εκεί το Συμβούλιο συμφώνησε να κινηθούμε προς μια κοινή προσπάθεια, μια κοινή βάση, ε, βάση περιπτώσει. για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ένα βήμα μόνο είναι αυτό βέβαια, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση για να το κάνουμε αυτό. Εγώ τι να κάνω, μόνο έκκληση μπορώ να απευθύνω, να παροτρύνω, να ενθαρρύνω τους υπουργούς. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της ομάδας εργασίας, να καλέσουμε ε, τους εμπειρογνώμονες, να συζητήσουμε και με το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να δημορφωθεί έτσι το χρονοδιάγραμμα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με εμπειρογνώμονες, με συζητήσεις και στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, το ΚΟΡΕΠΕΡ. Όλα αυτά χρειαζόμαστε. Αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είπα και στον κύριο Λίζε ότι είμαι διατεθειμένος να δω τις δικές σας προτάσεις, να τις εξετάσω και να βολιδοσκοπήσω τους υπουργούς. Τώρα, αν με ρωτάτε συγκεκριμένα αν μπορούμε τον Νοέμβριο ήδη να έχουμε καταλήξει, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Να τα ξαναπούμε αν θέλετε τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο για να δούμε πώς θα έχει μέχρι τότε το τοπίο. Εγώ είμαι χειρουργός και ιστορικός ταυτόχρονα και έχω συνηθίσει να ε, λειτουργώ με συγκεκριμένο τρόπο, με ακρίβεια και με στόχους ε, ρεαλιστικούς. Κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας έγιναν κάποιες πρόοδοι. Τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς. Πάντα σε διάλογο μαζί σας. Περιγράφοντας ε, ένα πραγματικό πρόγραμμα, μια ημερήσια διάταξη με ενδιάμεσα στάδια όπου θα αξιολογούμε κάθε φορά τα επιτεύγματα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέποντας και κάνοντας πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε και τι κάνουν και οι κυβερνήσεις. Να τις παροτρύνουμε ακριβώς να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες. Έτσι απαντώ στον Πέτερ Λίζε. Και ε, στην ερώτηση της κυρίας Ροτ Μπέρντ, θέλω να τονίσω και πάλι ότι ε, έχουμε τέσσερις μήνες μόνο στη διάθεσή μας για τη Λίντα Μακάβαν. Ε, μα ρωτήσατε για την οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Είμαι μεταξύ κυρίων. που θέλουν να υποστηρίξουν την ειλικρίνεια. Το είπε και ο κύριος ε, Σλίτερ για τις δραστηριότητες των ομάδων πίεσης, των λόμπι. Και με ενδιαφέρει πολύ και το θέμα της διαφάνειας. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες, ισχυρίζονται ορισμένοι, για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εγώ ως γιατρός μπορώ να σας πω ότι έτσι μακρινόμαστε από τη λύση του προβλήματος. Δεν είναι το σωστό ερώτημα αυτό. Το θέμα είναι αν ε, βλάπτει την υγεία το κάπνισμα. Ναι ή ου. Στον τριμερή διάλογο θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει το Δεκέμβριο αυτό. Είναι πολύ σημαντικός στόχος, διότι, γενικότερα διότι το κάπνισμα και ε, η κατανάλωση προϊόντων καπνού είναι κάτι που βλάπτει την υγεία. Είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Ε, εδώ και 200 χρόνια είμαστε όμοιροι της καπνοβιομηχανίας που μας έχει κάνει να καπνίζουμε. Το ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, το ξέρω ότι υπάρχει και θέμα ε, εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία και ότι δεν θα πρέπει να καταστραφεί. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά και όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου γύρω από αυτό το θέμα κατανοούμε όλη την επιχειρηματολογία και τον τρόπο με τον οποίο ε, δρά το Συμβούλιο. Όπως και να έχουν τα πράγματα όμως θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια προόδου και ο τριμερής διάλογος να ε, εκπονήσει θέσεις θεραλές και πρέπει να σας πω ότι έχω όραμα και πρέπει να έχουμε οράματα και όνειρα στη ζωή μας αν θέλουμε να βάζουμε στόχους και να πετυχαίνουμε κάποια πράγματα. για τις κλινικές δοκιμές τουλάχιστον στο Συμβούλιο θα ε, μπορούσαμε να εκπονήσουμε μια κοινή θέση, μια πρώτη ε, αφετηρία για να συνεννοηθούμε ε, και να έχει επιτύχει και η Προεδρία μας. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα μπορούσαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα Έχουμε αυτή την ημερήσια διάταξη, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, προφανώς ε, θα το ξαναπούμε. Θα ε, το ξανασυζητήσουμε. Ως χειρουργός, σας είπα, δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο, δεν έχω πρόβλημα, ε, δεν φοβάμαι τη σκληρή δουλειά. Συμφωνώ με τον κύριο Λίζε που είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, να την ολοκληρώσουμε και να μην διονύζεται αυτό το θέμα. για την ε, ε, οδηγία για τα προϊόντα καπνού και τα ιατροτεχνολογικά. Και ο κύριος Λίζε και η κυρία Ροτ Μπέρεν ρώτησαν αυτά τα θέματα και το χρονισμό. Είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όμως και στα χρονοδιαγράμματά μας και στους στόχους μας και σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, να τα κοιτάμε αυτά τα θέματα τον Οκτώβριο για ε, τα πειράματα, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για τις διαγνωστικές μεθόδους in vitro και μετά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα είμαστε σε θέση να πούμε εάν ε, πετύχαμε κάτι χειροπιαστό ή όχι. Και θα σας παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα και για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Μιλήσατε για το πρόβλημα μετανάστευσης υγειονομικού προσωπικού ε, γιατρών και νοσηλευτών. Θα πρέπει να δούμε και το κοινωνικό, και το κοινωνικό dumping που υπάρχει. Όλα αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη ε, όταν συζητούμε για την αηφορία των συστημάτων. Τα συστήματα των κρατών μελών ε, δεν είναι όλα στην ίδια κατάσταση αλλά στο σχέδιο των συμπερασμάτων θα ασχοληθούμε όλα, με όλα αυτά τα θέματα. Και με το φω. Και η διάσκεψη των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Βίλνιους ασχολείται με αυτά τα θέματα. Η αηφορία των συστημάτων υγείας έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Με τη διαμόρφωση των τιμών, με την αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εγκαταστάσεων και σε αυτή την άτυπη συνάντηση στο Συμβούλιο που σας είπα αποφασίσαμε να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή στην ελόγω διάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις σημαντικότερες θέσεις, τα συμπεράσματα και ε, στη συνέχεια θα ε, ασχοληθεί και με την αηφορία και την βιωσιμότητα των συστημάτων. Όλα αυτά είναι σημαντικά για το μέλλον, για το επόμενο διάστημα, πολύ δε περισσότερο που τον Οκτώβριο θα πρέπει να εφαρμοστεί οδηγία για την παροχή υπηρεσιών, τη διασυνοριακή. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη χρηματοδότηση και με τη στελέχωση Πολλοί οι τομείς λοιπόν που ε, ε, έχουν επιπτώσει στην αηφορία των συστημάτων υγείας. Σε σχέση με όλα αυτά υπάρχει και το ζήτημα του κανονισμού για τα τέλη ε, που καταβάλουν οι εταιρείε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την έγκριση των φαρμάκων τους και εκεί μπορούμε να έχουμε πρόοδο στο Συμβούλιο. Δεν είναι τόσο επίμαχο αυτό το θέμα, ξέρετε, μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αηφορία των συστημάτων, σας είπα, και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση. Συνοψίζω, για να τελειώσω, λέγοντας ότι Όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλα. Είναι μια δέσμη. Ελπίζω στο μέλλον να μπορέσουμε από κοινού πάντα και σε συνεργασία να προωθήσουμε αυτά τα θέματα και να καθορίσουμε τους στόχους μας. Ελπίζω το Συμβούλιο να αντιδράσει θετικά να αξιολογήσει θετικά αυτούς τους στόχους, ιδιαίτερα για την οδηγία καπνού. Που είναι ένα ιδιαίτερο κοινό εγχείρημα. Και βεβαίως περιμένουμε το φινόπορο μια θετική έκβαση στην ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Υπολογίζουμε σε εσά και ελπίζουμε να δοθεί η διαπραγματευτική εντολή και γιατί όχι μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αρχίσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων. Για την κυρία Παρβάνοβα. Και τη διαφάνεια ε, στον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων. Προχτές το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών με ρώτησε το ίδιο ο Βέλγος υπουργό Υγείας. Και τα κράτη-μέλη μίλησαν, αλλά είχαν πάρα πολύ διστάμενες απόψεις. Ορισμένες χώρες θεωρούσαν ότι αυτό είναι αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα και δεν τίθηκαν αυτό το θέμα και γιατί ασχολούμαστε με αυτό. Έξι κράτη-μέλη μια συγκεκριμένη ομάδα κρατών, ενώ κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Άτυπο ήταν το Συμβούλιο. Θα μπορούσε να τα συζητήσει αυτά τα θέματα. Και συμφωνήσαμε να συζητηθεί αυτό το θέμα στην ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. και συμφωνήσαμε ότι θα, θα βοηθούσε πολύ μια τέτοια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου για αυτό το θέμα. Η κυρία Άννα Ρόσπαχ μίλησε για τη φυματίωση. Πρέπει να σας πω ότι με θλίψη και μεγάλη οδύνη είναι ε, κάτι που αντιμετωπίζουμε και είναι προβληματική η αντιμετώπιση της ε, φυματίωσης στα ε, πρώιμα στάδια. Υπολοιπόμεθα σε σχέση με αυτό. Το ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με την αντοχή στα αντιβιωτικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα κακής θεραπείας. Η φυματίωση δεν την χάνει πάντα τη σωστή θεραπείας. Δίνονται λάθο φάρμακα ή με λάθος τρόπο και έτσι αυξάνεται η αντοχή των μικροβίων στην, ε, στα αντιβιωτικά. Γιατί το τελευταίο διάστημα ο ασθενής δεν πηγαίνει στο γιατρό, πηγαίνει στο διαδίκτυο, στο Google και ψάχνει την ενημέρωση και ε, προχωρεί σε αυτοθεραπεία. Ε, αγοράζει μόνο στα φάρμακα. Γίνονται διάφορες προσπάθειες να καταρχηθεί η ιατρική περίθαλψη, ακόμα και ο εμβολιασμό και θέλουν οι ασθενείς να είναι σε θέση να αυτοθεραπεύονται, να θεωρούν ότι μπορούν μόνοι τους να τρέχουν σε διάφορα φάρμακα θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ασθενείς ότι δεν, είναι δραματικά αυτά τα λάθη, είναι τραγικά. Η φυματίωση έχει και σχέση με την κατανάλωση νοπνεύματος, με τη φτώχεια και με πολλούς άλλους παράγοντες κοινωνικής φύσεως όμως. Και με άλλα νοσήματα. Οι ασθενείς δεν τηρούν τις οδηγίες των ιατρών, ούτε τη θεραπευτική αγωγή που τους χορηγείται. Εξού και η αντοχή μετά των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Αυτά θα πρέπει να τα συζητούμε στα διάφορα επιστημονικά φόρα και να αντιμετωπίζονται ως θέματα πρόληψης. Ε, και το θέμα αυτό δεν είναι επίκαιρο μόνο τώρα λόγω της Λιθουανικής Προεδρίας, είναι οξύτατο και θα μας συνοδεύει και τα επόμενα χρόνια. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορούμε να λύσουμε εμείς κατά τη διάρκεια ε, της Προεδρίας μας. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα και τα υποθέματα, γιατί όπως σας είπα έχουμε ένα τετράμινο. Ο συνάδελφος Γιούστας Παλέτσκης μίλησε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και αναφέρθηκε σε πρότυπα και προδιαγραφές. Όντως, για η φορεία και βιωσιμότητα των συστημάτων ε, υγείας θα πρέπει να ε, συνδέεται με την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία. Δηλαδή, τα συστήματα δημόσιας υγείας θα πρέπει να ανοίξουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, πλουσίους και φτωχούς. Και σε σχέση με αυτό λοιπόν και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και θα δούμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη βιωσιμότητα των συστημάτων. Έτσι νομίζω θα έρθουν οι ανισότητες και θα παρακαυθούν ή θα καταργηθούν. Υπάρχουν πολλά μέσα στη διάθεσή μας για να υλοποιηθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Με τον κύριο Βιτόριο Πρόντι. Σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ ως Ευρωπαίος και μέλος της συντακτικής συνέλευσης Είμαι υπέρ της υποχρεωτικής ισχύω ε, του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πετύχει ήδη πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Το 1982 συνελήφθη και φυλακίστηκα. Και τότε για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όνειρο και μόνο. Και σήμερα πιστέψτε με, δεν το έχω πιστέψει ακόμα ότι είμαι προεδρεύων. Ε, τέτοια τεράστια αλλαγή κατάφερα να, τα, να τη ζήσω κατά τη διάρκεια της σύντομης ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό. Για την υγεία για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, για την ίση αμοιβή για ίδια εργασία και στον τομέα της υγείας. Αυτά είναι καθημερινά προβλήματα και ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα πρέπει να φροντίσουμε, να αγωνιστούμε και να πούμε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου πραγματικά εφαρμόζονται στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να κάνουμε και εδώ πρόοδο. Λοιπόν, με ρωτήσατε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Προσωπικά φρονώ ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι μια απόπειρα να συνεχιστεί το κάπνισμα και αυτή η μπίζνα γύρω από τον καπνό με άλλο τρόπο. Οικονομική δραστηριότητα. Προσωπική άποψη. Θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει φαρμακευτικό προϊόν, αλλά εγώ που είμαι γιατρός δεν το θεωρώ φάρμακο. Αυτό είναι άλλη μία εξάρτηση και τίποτα άλλο. Και πολλοί γιατροί θα αγωνιστούν έτσι ώστε αυτή η νέα ασθένεια να αντιμετωπιστεί και να ε, ιαθεί. Ε, αναφερθήκατε στο διαδίκτυο. Γιατί εκεί πωλείται τώρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πριν από λίγο καιρό μου τηλεφώνησε ο πατέρας μου και μου ζήτησε, όχι δικός μου, ένας πατέρας, και μου ζήτησε βοήθεια ε, γιατί ο γιος του αγοράζει ηλεκτρονικά τσιγάρα από το διαδίκτυο. Και με ρώτησε γιατρέ, τι τσιγάρο είναι αυτό. είναι μια νέα μάστιγα και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να εθελοτυφλούμε σαν να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Για την κυρία Μαρκουνάιτε, η οποία μίλησε για την εκπαίδευση, για την ενημέρωση της κοινωνίας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα ενημέρωση στα διάφορα κράτη-μέλη. Διαφέρει αυτό από χώρα σε χώρα και η κάθε πρόοδος διαφέρει. Υπάρχουν χώρες που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικές, διστακτικές και προτείναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μεταφερθεί ε, αυτή η προσπάθεια και να ανταλλάξουμε εμπειρίες που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάλι να συντονίζονται τα κράτη-μέλη για να υπάρχει ενημέρωση από τον τύπο. Και μπορούμε έτσι να επηρεάσουμε τις συμπεριφορές των νέων. Από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση από διάφορα μέσα ενημέρωσης κάθε φορά και τον τύπο ε, στην εκάστοτε χώρα θα μπορούσαμε να ενημερώνουμε τον πληθυσμό και για θέματα δημόσιας υγείας. Η κυρία Μόρκουνάιτε μίλησε για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπως είναι Αλτσχάιμερ και άλλες νόσοι η ψυχική υγεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ένα θέμα το οποίο αφορά και αυτή την αρρώστια με τον α ή β τρόπο. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, κάποια εγκεφαλικά επεισόδια, ε, συνδέονται και με την ψυχική υγεία. Στη διάσκεψη για την ψυχική υγεία στο Βίλνιους θα ασχοληθούμε και με αυτά τα επιμέρους στοιχεία των νοσημάτων αυτών. Και αυτό έχει σημασία για τα συστήματα υγείας. Για να δούμε λοιπόν ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες επιπλέον προκλήσεις. τίθενται και κοινωνικά ζητήματα. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα θα πρέπει να εντάσσονται στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας, να είναι πιο εύκολη η ζωή τους για να μειωθούν και τα κρούσματα των αυτοκτονιών. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολύ εύθραυστοι, πάρα πολύ ευαίσθητοι. Αν δεν έχουν αρκετό εισόδημα, αν δεν έχουν αρκετή σύνταξη, αν δεν έχουν ε, ίδιους πόρους. Απελπίζονται. Καταλαβαίνετε όλα αυτά τα προβλήματα είναι σε ένα συνολικό πλαίσιο και συνδέονται μεταξύ τους. Οι Υπουργοί Υγείας λοιπόν είναι εκείνοι που καλούνται να απαντήσουν και μπορούν να το κάνουν αυτό και να διατρανώσουν ότι είναι μια πολυτομεακή προσέγγιση. Και αυτή θα δώσει την απάντηση και σε αυτά τα ζητήματα που με ρωτήσατε και που τίθενται για ανθρώπους ε, ψυχικά νοσήματα, με ψυχική, διανοητική ή σωματική αναπηρία. Έτσι χρειάζεται μια ευρύτερη προσέγγιση και σε σχέση με αυτά να είναι αντίστοιχη και η χρηματοδότηση από τον ένα κλάδο στον άλλον. για να απαντήσω και στην άθελφο από την Κροατία, την κυρία Γκόρσαν. Σας καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή και τη χώρα σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια. Ο Υπουργός Υγείας σας ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ο νέος επίτροπος είναι πάρα πολύ δραστήριος και του είπα ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ στενά. Αναφερθήκατε σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό ε, μετά την ένταξή σας. Όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά θέλω να σας πω εδώ σε αυτή τη φιλική ομίγυρη ε, ένα αστείο, μου επιτρέπετε. τρομάζουμε τόσο πολύ τον κόσμο. Θυμάστε την ιστορία του Πολωνού Ιδραυλικού. Κάποια στιγμή μετά την ένταξη κυκλοφόρησε η φωτογραφία, μάλλον δημιουργήθηκε αυτό, αυτή η εικόνα του Πολωνού Ιδραυλικού που είναι ο μέγας κίνδυνος για την Ευρώπη ολόκληρη και θα μας κατακλείσει. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες τη διαμόρφωση της εικόνας και της αντίληψης της κοινή γνώμης. Προβλήματα υπάρχουν, μπορούμε να τα συζητήσουμε, έχουμε εμπειρίες συλλέξει και από προηγούμενες ε, καταστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αηφορία και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας μας και σε σχέση με τα προβλήματα που έχουμε στα διάφορα κράτη-μέλη. από πού φεύγει το ιατρικό και το υγειονομικό προσωπικό. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά και δεν θα πρέπει να μας τρομάζουν. Είμαι αισιόδοξο και μπορώ να σας πω ότι τίνουμε χείρα βοηθείας, αν χρειάζεστε. Και στην Κροατία θα είμαστε στο πλευρό σας. Ελπίζω να απάντησα σε πολλές ερωτήσεις. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να γίνω τέλειος συγκεκριμένος. Καμιά φορά δεν έχω και συγκεκριμένες απαντήσεις, γι' αυτό χρειάζομαι τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Υπουργέ. Νομίζω απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις και είναι σπάνιο να ακούει κανείς από Υπουργό ότι δεν έχω απάντηση σε όλα. Νομίζω απαντήσατε εκτενέστατα, αναλυτικότατα, απαντήσατε και σχολιάσατε κάθε τοποθέτηση και κάθε ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι δεν ζητεί κανείς άλλο το λόγο, οπότε ήταν ένας και μοναδικός ο γύρος των ερωτήσεων, τον οποίο καλύψατε. Σας εύχομαι και σε και στη χώρα σας για το έργο που σας περιμένει. Ε, καλή τύχη, καλή αντοχή, καλή δύναμη δεν μπορώ παρά να πω ότι η δική μας Επιτροπή θα είναι πάντα στο πλευρό σας με κριτικό πνεύμα και μάτι, αλλά προοδευτικό ξέρετε ότι είμαστε η μεγαλύτερη νομοθετική φύσεως Επιτροπή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάντα γνώμονά μας, μας είναι ε, το καλό των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Γιατί για την υγεία ο καθένας μια υγεία έχει και είναι το ύψιστο αγαθό όλων μας. Και αυτό θα πρέπει να το προωθούμε, να το προάγουμε, να το βελτιώνουμε και σε καιρού ισχνών αγελάδων και δημοσιονομικών στενοτήτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει τα μάλα η παρουσία σας εδώ. wir machen jetzt weiter. Hat jeder seine Abstimmkarte? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, την πήρατε την κάρτα ψηφοφορία σας για τις διακοπέ μην την αφήσετε εδώ. Καλές διακοπέ σε όλους. Ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία, για τις ερωτήσεις σας. Ε, φορτώστε τις μπαταρίες σας και τα ξαναλέμε τέλη Αυγούστου όλοι υγιείς και ε, με χαρά αρχές Σεπτεμβρίου. Γεια σας, καλές διακοπές.